ηλεκτρονικό μα ταχυδρομείο για μια ολόκληρη εβδομάδα. Θα ήθελα να ενημερωθώ λοιπόν πόσο σοβαρό ήταν ο κίνδυνο, αν ήταν μόνο προληπτικό το μέτρο και στη τελευταία ανάλυση πόσο ευάλωτο είναι το ηλεκτρονικό μα σύστημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα το επαληθεύσουμε και θα σα ενημερώσουμε. Thank you very much. Uh... Ε, η κυρία Γκίγιομ τώρα, η κυρία εισηγήτρια. Παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Πρόεδρε, ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Αυτή την εβδομάδα προχωρούμε στην πρώτη φάση αναθεώρηση τη ε, οδηγία για τι διαδικασίε. Την Τετάρτη θα λάβουμε θέση για την αναθεωρημένη πρόταση τη Επιτροπή για την κοινή διαδικασία σε ό,τι αφορά τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτο του πρόσφυγα. Η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου είναι ουσιαστική στον διάλογο που θα συνεχιστεί με το Συμβούλιο του επόμενου μήνε για ένα θέμα που πιστεύω ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πακέτο για το άσυλο και για το οποίο δυστυχώς ε, δεν προχωρούν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Θα αποτελέσει η βάση τη νέα εκδοχή τη οδηγία που ελπίζω ότι θα επιτρέψει να τηρήσουμε το 2012 ως στόχο δημιουργία του, Ευρωπαϊκού, του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Η ψηφοφορία για την έκθεση γίνεται τη στιγμή που τη αρμοστήρια του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια μεγάλη έρευνα για 44 βιομηχανικές χώρες που δείχνει ότι αντίθετα από τις ιδέες που υπάρχουν, ο αριθμός των αιτητών ασύλου μειώθηκε κατά 44% τα τελευταία 10 χρόνια και κατά 5% σε ένα χρόνο. Μια τέτοια, ε, μια τέτοια διαπίστωση μας οδηγεί στο να αναρωτηθούμε γιατί μειώθηκαν οι λόγοι αναχώρησης ή αυξήθηκαν οι αυστηροί έλεγχοι τη μετανάστευση σε κάποιε χώρε. Επίση, η έκθεση δείχνει ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε υφίστανται σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα τη ευθύνη στον τομέα του ασύλου, ενώ δεν έχουν κατά ανάγκη όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχουν κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τη και να αποκτήσει για τον σκοπό αυτό σαφεί κανόνε. Αυτό με οδηγεί στο ζήτημα, τη διαδικασία ασύλου για να υπενθυμίσω τα βασικά ζητήματα. Συχνά ε, χαρακτηρίζεται η οδηγία αυτή ως κατάργωση των χειρότερων εθνικών πρακτικών, αλλά έχει δύο βασικά προβλήματα. Δεν, προστατεύει επαρκώς τα δικαιώματα των ετούντων, ενώ υπάρχουν ε, αγνοεί τις τεράστιες ανισότητες αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις με το, μεταξύ των διαφέρων συστημάτων ασύλου στην Ευρώπη. Δύο παραδείγματα. Το ποσοστό θετικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό στα κράτη-μέλη το 2009 περνάει από το 65% σε κάτω από 1%. Οι προθεσμίες κατάθεσης προσφυγών κατά αρνητικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό ποικίλει από, το 2, από 2 έως 30 ημέρες. Οι ανισότητες λοιπόν είναι σημαντικές μεταξύ των κρατών μελών. Για τους λόγους της ε, ε, ταχύρυθμης διαδικασίας, της αποτελεσματικής προσφυγής, της προστασίας. Αυτό είναι ασύμβατο με ένα καθεστώς, ενιαίο καθεστώς αστήλου που πρέπει να παρέχει ισοδύναμη προστασία σε όλη την Ένωση. Επιπλέον έρχεται σε αντίφαση και με ένα από τους λόγους της, ε, του θέσπης του κανονισμού Δουβλήμου 2 που, προβλέπει, που υποθέτει, που θεωρεί ως αυτονόητο ότι είναι ισοδύναμα ε, ε, τα καθεστώτα ασύλου στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει δίκαιε, προσπελάσιμε, ασφαλεί και αποτελεσματικέ διαδικασίε ασύλου. Θα ήθελα εκ νέου να απαντήσω σε κάποιες δηλώσεις των κατηγόρων του κειμένου αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι παράλογες. Αυτοί λένε ότι η οδηγία στην ουσία περιλαμβάνει απλά αύξηση του κόστους. Οι αλλαγές θα οδηγήσουν όντως σε βραχυπρόθεσμες αυξήσεις του κόστους. Αλλά ας είμαστε λίγο πιο ε, ξεκάθαροι. Η κακή διαδικασία. Η ανεπαρκής ασφάλεια κοστίζει αυτή τη στιγμή πολύ στα κράτη-μέλη. Δύο στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω. Ο μεγάλος αριθμός προσφυγών και η διάρκεια των διαδικασιών που δημιουργούνται από αυτό. Πρέπει να φύγουμε από μια μανιχαϊστική αντίληψη του ασύλου που μιλούν ότι το άσυλο είναι μόνο κατά ότι χρησιμοποιείται, ε, κάποιοι χρησιμοποιούν το άσυλο, το, το να χρησιμοποιούμε την μετανάστευση για να καταπολεμήσουμε το, το άσυλο είναι λάθος. Δείτε τι γίνεται στην, στις αραβικές χώρες. Είναι ευθύνη της Ένωσης να δώσει μια δίκαιη προστασία στα θύματα διώξεων. Υποστηρίζω λοιπόν την προσέγγιση της Επιστροπής για την βελτίωση των διαδικασιών σε πρώτο βαθμό, το front loading, διότι μια απόφαση ποιοτική σε πρώτο βαθμό θα είναι θετική και για τα θύματα διώξεων, αλλά θα επιτρέψει στέρεες αποφάσεις στις αρμόδιες αρχές με βελτίωση της αιτιολόγησης των αποφάσεων και μείωση των κινδύνων ακυρώσεως των αποφάσεων αυτών, να εντοπίζει καλύτερα τις ε, καταχρηστικές ή αβάσιμες ε, προσφυγετήσεις και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην αναχώρηση των πραγματικά απορριφθέντων αιτητών. Δύο λόγια για τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Το δικαίωμα σε δωρεάν νομική συνδρομή σε πρώτο βαθμό, κατά την άποψή μου, αποτελεί βασική εγγύηση για τη βελτίωση τη ποιότητα των αποφάσεων. Μια καλύτερη λήψη υπόψη των ευάλωτων ομάδων, για τις οποίες η σημερινή οδηγία σιωπεί. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Επτά λεπτά έχετε συνολικά. Θέλετε να τα κόψετε πέντε-δύο. Θα συνεχίσω, λέει ο μιλήτη. Μισό λεπτό ακόμα. Τρίτο ζήτημα οι φιλόδοξε προθεσμίε ε, προσφυγή που περιορίζουν το δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή και η σημαντική αύξηση των, ε, των ταχύρυθμων διαδικασιών. Αλλά για το ζήτημα της ασφαλούς χώρας ζητούμε κοινή ε, εμφάνιση κοινή κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο με συναπόφαση. Συνολικά, η τελική έγκριση της έκθεσης θα πρέπει να αποτελήσει ένα σοβαρό μήνυμα του Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Οι κόκκινες γραμμές του Κοινοβουλίου έχουν τεθεί πολύ κοντά στην εναρμόνιση προς τα άνω των προτύπων προστασίας. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι όλοι κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο. Και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Σασίλια Μάστρομ. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Συγκητρία, είναι πολύ σημαντική η ψηφοφορία για το θέμα του ασύλου αυτή την εβδομάδα γιατί θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ολοκλήρωση της δεύτερης ε, φάσης ενός κοινού συστήματος για το άσυλο για το 2012 ε, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρόγραμμα μέσα στο πρόγραμμα Στοκχόλμης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκυγιόμ ιδιαίτερα για την ε, αποφασιστική της δέσμευση και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει. Έχει επιδείξει μεγάλη επιμονή και υπομονή και κατανόηση των αναγκών των ετούντων το άσυλο καθώ και των προκλήσεων που αντιμετωπίσουν οι αρχέ των κρατών μελών. Η νέα λοιπόν διαδικασία αυτή για την ε, χορήγηση του ασύλου θα αποτελέσει την ε, θεμέλιο, το θεμέλιο λίθο για ένα κοινό σύστημα ασύλου. Όπω είπατε και εσεί, κυρία Κιγιόμ, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα ασύλου οπουδήποτε και αν κατατίθεται η αίτηση για την χορήγηση ασύλου. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικέ διαδικασίε, πράγμα το οποίο βεβαίω δεν είναι κατανόητο μέσα στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ίδιε ισχύουσε διεθνεί συμβάσει και με τι ίδιε ισχύουσε ευρωπαϊκέ αρχέ, γιατί να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα δίκαιο, αποτελεσματικό, που να μην επιτρέπει καταστράτηγηση του συστήματο, αλλά και να εξασφαλίσει ταυτόχρονα σεβασμό και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όμω εάν υπάρχουν κοινοί κανόνε οι οποίοι θα εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο Τη προστασία ε, και του τρόπου λήψη αποφάσεων από τις αρχές ε, ε, για την έγκριση του ασύλου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω αρχή. Αυτό από ό,τι βλέπουμε υποστηρίζει και η κυρία Γκυγιόμ και η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών εν γέννη. Πολλέ είναι οι τροπολογίε στο σχέδιο τη εκθέσεως που ενισχύουν ιδιαίτερο στο επίπεδο των εγγύσεων για τον ετούντα το άσυλο και ιδιαίτερα για του ανηλίκου. Ορισμένε εκ των τροπολογιών επίση στόχο έχουν εξασφαλίσει περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και εισάγουν ε, κάποιου επιπλέον λόγου για αναγνώριση ταχύρυθμη διαδικασία. Η έννοια τη περιγραφή τη τρίτη χώρα πιστεύω ότι είναι πολύ φιλόδοξη. Ε, Επίση, κατά περιγράφονται εκ νέου οι ορισμένοι κανόνε και καταγράφονται εκ νέου οι πρακτικέ που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι με την ε, ε, λύση που προτείνει η κυρία Γκυγιόμ μπορούμε να, δώσουμε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νομικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι ε, έχουμε προσπαθήσει να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τι προτάσει αυτέ που έχουμε καταθέσει και πιστεύω ότι η ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσει σημείο κάμπη. Με πολύ μεγάλη προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει και θα μελετήσει τι δικέ σα τροπολογίε όπω θα εγκριθούν και θα συνεργαστούμε από εδώ και μπρο πάλι μαζί σα στενά για την ε, περαιτέρω πορεία αυτή τη προτάσεω. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε. Στη συνέχεια η κυρία Μόνικα Χολμάια, εξ του ΕΛΚ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, καταρχήν Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά για τις πολλές επαφές και συζητήσεις που είχαμε με την εισηγήτρια αλλά επίσης και με την Επίτροπο και τους κοιόδης εισηγητές. Και σε κάποιους τομείς καταφέραμε να πετύχουμε καλούς συμβιβασμούς. Όπως ανέφερε μόλις η Επίτροπος Μάλμστρομ, ανήκει και αυτό σε αυτό το πλαίσιο και ο συμβιβασμός ε, για την συνδρομή όσον αφορά το κόστος ε, για την παροχή υπηρεσιών και προστασία των ανηλίκων και ιδιαίτερα των ευάλωτων ατόμων που και για τη γλώσσα καταφέραμε να βρούμε ένα λογικό συμβιβασμό καθώς επίσης και για το θέμα των ασφαλών τρίτων κρατών επίσης συμβιβασμό. Στόχος είναι καταρχήν οι διοικητικές διαδικασίες ε, να βελτιωθούν όσον αφορά την ποιότητά του, να αναβαθμιστούν ώστε οι ετούντε άσυλο οι οποίοι διώκονται να μπορούν το δυνατόν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά να την χάνουν συνδρομή και βοήθεια. Είμαι απόλυτα υπέρ του ότι να υπάρχουν ανάλογα ελάχιστα όρια, προδιαγραφέ δηλαδή στα κράτη-μέλη. Στο κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε επιμέρου τροπολογίε που στοχεύουν να τροποποιήσουν το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Πολλέ φορέ οι καλέ προθέσει μετατρέπονται στο αντίθετο. Πολλέ φορέ ε, υπάρχουν ε, διαδικασίε που επιβραδύνουν ε, το, την συνολική διαδικασία και καταχρηστικά κιόλα. Και θα αναφέρω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, ένα ετών άσυλο μπορεί τρει φορέ ε, να θέτει ένα τέτοιο αίτημα και έχει ε, απέτηση, μπορεί να έχει απέτηση τρει φορέ για την εξέτασή του. Τώρα, για την μη επιτάχυνση μια διαδικασία όταν κάποιο δεν αναγνωρίζεται ω πρόσφυγα υπό την σύμβαση τη Γενέβη για ε, παράδειγμα σε σχέση και με την Τινησία και άλλες περιπτώσεις. Χωρίς, ε, υπάρχουν τροπολογίες ε, που χωρίς να αναφέρονται σε κάποιο ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός αναφέρονται σε αυτή την πτυχή. Επίσης όσον αφορά την αρνητική έκβαση ενός αιτήματος ετούντος άσυλο θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη υπογραφή για το αίτημα αυτό από τους αρμόδιους όταν παίρνει, αναμένει κάποιος μια αρνητική τέτοια απόφαση μόνο θα μπορούσε να αρνηθεί την, ε, την παραλαβή του ταχυδρομείου ή του μηνύματος αυτού Ευχαριστώ κυρία. Ο κύριο Κλοντ Μωράης στη συνέχεια παρακαλώ από πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Πρόεδρε, Λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματο ε, της Σοσιαλιστικής Ομάδας λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη πραγματικά κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη κάνουν λόγο για την ολοκλήρωση ενός πακέτου για το άσυλο από το 1999 και αν υπάρχει κάποια επιταγή να προχωρήσουμε, πραγματικά αυτή είναι σήμερα με την κρίση στη Βόρεια Αφρική και στην ε, Μεσόγειο. Και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πρακτική και λογική πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Η κυρία Γκυγιόμ συνεργαζόμενοι όπως είπαμε με όλους τους σκιώδεις εισηγητές εξεπώνησε μια πρόταση που είναι λογική, ευαίσθητη, αποτελεσματική και δίνει τον ακρογωνιαίο λίθο για το πακέτο για τα μέτρα ασύλου σε σχέση με την κοινότητα. Γι' αυτό είναι τεράστια σημασία σε αυτό. Αν μπορούμε να επαναλάβουμε την πλειοψηφία που σημειώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πακέτο για το άσυλο που θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ανησυχίες και τα μελήματα των μελών. Να δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Είχα ασχοληθεί με πολλές τέτοιες περιπτώσεις ως δικηγόρος για τους ετούντες άσυλο και ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει μια ταχεία, λογική και δίκαια διαδικασία και όταν έχουμε την περίπτωση του front loading, το γεγονός ότι ε, σε σχέση με την ποιότητα της λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά κράτη-μέλη οδηγεί αυτή η κατάσταση όσο έχει σήμερα σε υψηλό κόστος. Κάνουν λόγο λοιπόν για χρηματοοικονομικές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως ε, ότι η ποιότητα η οποία θα αναβαθμιστεί θα διασφαλίζει ότι θα λειτουργούν σωστά οι διαδικασίες. Εκεί θα εξοικονομούμε κονδύλια, θα είμαστε δίκαιοι και θα δρούμε γοργά. Και σε σχέση με αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δικαιοσύνη, δίκαια, ε, η ανάγκη να είμαστε δίκαιοι μέσα σε ένα εύλογο πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα επίμαχα θέματα. Επίσης ε, θα πρέπει να τονιστεί ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να διεξάγεται μόνο για το κόστος ε, για την εναρμόνιση αυτών των ε, μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε τέτοιου είδους λοτερία για τα θέματα ασύλου δεν θα δίνουμε προσοχή στην πραγματικότητα της αύξησης κιόλας των ετούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βρισκόμαστε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση οι κανονισμοί σε σχέση με τις διαδικασίες αφορούν ίσως το πιο περίπλοκο μέρος ε, για το πακέτο για τα μέτρα για τους ετούντες ε, άσυλο και το άσυλο γενικά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ευθύνες μας και να υπομισθούμε τις ευθύνες αυτές όταν έχουμε ανθρώπους που ε, στοιχίζονται και αναμένουν στα σύνορά μας. Γι' αυτό σε σχέση με τους σιώδεις εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν θέλω να ευχαριστήσω. Ας επαναλάβουμε το θετικό αποτέλεσμα που είχαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ψηφίζοντας και να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι είμαστε σοβαροί στο Ευρωκοινοβούλιο θέλοντας να ολοκληρώσουμε ένα πακέτο για τα θέματα ασύλου που θα είναι ευρωπαϊκό πλέον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίασή σας κύριε Μωράης και τώρα η κυρία Νάντια Χίρσα από Φιλελεύθερους και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καταρχήν ευχαριστώ θερμά την εισηγήτρια και τους εισηγητές. Είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις που κάναμε και στο τέλος νομίζω καταλήξαμε και σε καλούς θετικούς συμβιβασμούς. Παρότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ήταν όλα απλά, οι διαδικασίες δεν ήταν απλές. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι εμείς πάντα ακόμα υπερασπίζουμε το στόχο ότι το 2012 θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό, κοινοτικό ευρωπαϊκό σύστημα για το άσυλο. Και έτσι λοιπόν εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός, ώστε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο, ότι αυτό τον στόχο δεν τον έχουμε απεμπολίσει, δεν τον χάσαμε από μπροστά μας και ότι φυσικά θα δώσουμε συνέχεια. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο βέβαια, αλλά πρέπει να δείξουμε με σαφήνεια ότι το επιθυμούμε αυτό, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και θέλουμε να επιτευχθεί ένα κοινό σύστημα για το άσυλο. Δεν μπορεί να είναι θέμα τύχης μια λοτερία όταν κάποιος θέτει ένα αίτημα ε, ασύλου και η έκβαση, του είναι, ε, η έκβαση αυτού του αιτήματος είναι αβέβαια. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε κράτος μέλος να υπάρχει ένα ξεχωριστός, να υπάρχει ένα ξεχωριστός κατάλογος για το τι είναι ασφαλή τρίτα κράτη. Ή ένα κράτος, τρίτο κράτος είναι ασφαλές ή όχι. Και πρέπει αυτά ενιαία να αντιμετωπίζονται. Και πρέπει ατομικά να εξετάζεται για τον ετούντα άσυλο πραγματικά αν αυτό το κράτος είναι ασφαλές ή όχι ή αν σε μια ξεχωριστή ατομική κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα να αποφανθεί κανείς ε, και είμαι πεπισμένοι ότι στο τέλος τέλος θα αποκομίσουν κέρδος από αυτό, όφελος στα κράτη-μέλη. Και τώρα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά με ένα δίκαιο τρόπο με τα ταχύτερες διαδικασίες να προχωρούμε στην, στις αποφάσεις και στην έκβαση αυτών των αιτήσεων. Είναι αυτό νομίζω ένα δικαίωμα. Είναι δικαίωμα το άσυλο. Δεν είναι δώρο, δεν είναι χάρη που κάνουμε και πρέπει να έχουμε μια σαφή διαδικασία που θα διέπει τα θέματα ασύλου. Το χαιρετίζω το καταφέραμε εδώ για τους ανήλικους ε, να διευρύνουμε τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται για αυτούς. Υποστηρίζει η φιλελεύθερη ομάδα αυτό το, αυτό το στόχο στόχο και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αίσιο τέλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φλότρο. Φλότρο, παρακαλώ. Από τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έργο που έγινε για την έκθεση αυτή υπό την καθοδήγη τη κυρία Γκυγιών είναι πολύ σημαντικό. Το είπε η κυρία Μάλστρομ, είναι ο ακρογωνίο λήθο του Ευρωπαϊκού Σύστήματο Ασύλου. Και μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και του ευρωπαϊκού συστήματος υπάρχει ολόκληρο κενό τεράστιο ρήγμα στο οποίο βουλιάζουν και τα δικαιώματα των αιτητών και το σύστημα προστασίας στην Ευρώπη. Όταν έχουμε κράτη όπου οι θετικές απαντήσεις σε πρώτο βαθμό περνούν από το 1 στο 65%. Όταν σε χώρες όπως τη Γαλλία το 75% της προστασίας που χορηγείται σε Κωσοβάρους ε, και Αλβανούς δόθηκε ε, με προσφυγή και γνωρίζουμε ότι η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και το Συμβούλιο κατά συνέπεια θα πρέπει να ε, σπεύσει να εξετάσει την επιλογή που προτείνει η Επιτροπή και που ενισχύει η ποιότητα της έκθεσης της κυρίας Γκυγιόμ, δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, θα καταλάβαινε το Συμβούλιο ότι αυτό είναι θεμελιώδες. Τα κράτη που φωνάζουν δεν πληρώνουν, ούτε είναι και τα πιο φιλόξενα. Θα πρέπει να δούμε ότι σε σχέση με τον πληθυσμό η Κύπρος, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο είναι οι χώρες που έχουν περισσότερους και αυτοί μπορεί να μας πούν ποιοι είναι οι καλύτεροι κανόνες διεθνούς προστασίας των αιτητών ασύλου. Ευχαριστώ. Κύριε Φλότρ. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Χαίρομαι, Πρόεδρε, που γίνεται σήμερα η συζήτηση δεδομένη της, ε, ενόψη της ε, ψηφοφορίας ε, την Τετάρτη. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με τις παραγωγικές διαδικασίες να υλοποιήσουμε το στόχο μας για ένα ευρωπαϊκό σύστημα σύλλου το 2012 λαμβάνοντας υπόψη το έργο που κάναμε για το ζήτημα αυτό όλοι και γνωρίζοντας το πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος μπροστά, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κυγιόμ για την εξαιρετική δουλειά της και την ε, συνδιαλλαγή με την οποία αντιμετώπισε τις προτάσεις. Μπόρεσαμε έτσι να βελτιώσαμε σημαντικά τις διαδικασίες σε σχέση με τις διαδικασίες ασύλου στην Ένωση σήμερα, που ποικίλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Να σας δώσω κάποιες από τις νέες διατάξεις. Εξασφαλίζουμε ότι κάθε τιτής έχει τα επαρκή μέτρα μέσα για να τεκμηριώσει την αίτησή του και να πετύχει μία απόφαση μέσα σε 6 μήνες, όπως προσωπική συνέντευξη, δωρεάν νομική συνδρομή και παροχή των ε, αναγκαίων ε, δικονομικών εγγράφων. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ο κύριος Μπάτεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η υφιστάμενη οδηγία του 2005 για την διεθνή προστασία αναδιατυπώνεται ως οδηγία ως οδηγία υποδοχής όπως και η οδηγία υποδοχής που είναι εξέλιξη της κοινή πολιτική ασύλου και μετανάστευση τη Ένωση, όπω την θέτει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Η νέα οδηγία έχει η πρόθεση να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα για τα, που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια ε, εισόδου και αναγνώριση καθεστώτο πρόσφυγα και του όρου αναγνώριση. Έχει στόχο να εναρμονίσει την πολιτική ασύλου των κρατών μελών και να δώσει περισσότερα δικαιώματα και προνόμια σε αυτού που ζητούν άσυλο. Η παρούσα εισρωή πληθυσμών από τη Βόρεια Αφρική είναι άλλη μια ευκαιρία που δίνει στην Ένωση ε, την, ακόμα μια ευκαιρία να επεκτείνει τις αρμοδιότητές της. Η πολιτική ασύλου και μετανάστευση πρέπει να είναι κυρίαρχο δικαίωμα των κυρίαρχων εξαρτήτων κρατών. Η πρόταση οδηγίας κάνει, δείχνει ότι η συνδίκη της Λαβώνας κάνει αυτό ακριβώς που έλεγαν αντίπαλοι του ότι θα κάνει και γι' αυτό το λόγο δεν αφήσατε να γίνει και δημοψήφισμα σχετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στούπ. Πρόεδρε, το κόμμα μου... Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το κόμμα μου πάντα ήταν απόλυτα σαφές, κάθετα σαφές κατά της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ε, το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στην Ολλανδία είναι το καλύτερο που είχαμε. Έχει μια πολύ καλή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο στην ε, Ολλανδία. Τα κράτη-μέλη τέλεια μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα πλαίσια σε σχέση με τις ανάγκες ε, για το άσυλο. Αυτό το δικαίωμα, όπως το αποκαλούμε για το άσυλο, δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο βαθμό μετανάστευσης ε, για ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο κράτος ε, για να ζήσουν σε αυτό. Δείτε τι γίνεται στην Ιταλία, δείτε τι συμβαίνει στην Λαμπεντούζα εγκληματίες ε, οι οποίοι προσποιούνται ότι ε, ε, διώκονται και ζητούν άσυλο καταλήγουν εκεί είναι άτομα τα οποία είναι ανεπιθύμητα στην Ευρώπη. Η πολιτική μας είναι η πολιτική του να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση στα ίδια τα κράτη-μέλη μας αυτοί, αυτές οι αραβικές χώρες, οι μουσουλμανικές χώρες να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα που έχουν και όχι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους. Έτσι λοιπόν η πρόσβαση σε σχέση με ε, άτομα που προέρχονται από βάρβαρες χώρες με, βάρβα, με πολιτισμό βαρβαρότητας δεν θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην Ευρώπη. Διαδικαστικό εσείς. Ο συνάδελφος μόλις έκανε λόγο για ορδές βαρβάρων που προσέρχονται στην Ευρώπη, Πρόεδρε. Αυτή η κοινική τοποθέτηση δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς να υπάρξει κάποιο αντεπιχείρημα από πλευράς μας. Παρακαλώ αυτό να επισημαθεί και να ληφθεί υπόψη. Έχετε δίκιο. Θα καταχωρηθεί αυτό στα πρακτικά και σας ευχαριστώ για αυτή την παρατήρησή σας. Ευχαριστώ, συνάδελφε. ναι, παρακαλώ εσείς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα αν επιτρέπετε να διορθώσω κάτι, δεν είπα ακριβώς αυτό για ορδές βαρβάρων. Έκανα λόγο για ε, μια ε, περιοχή βαρβάρων. Δεν ήθελα να αναφερθώ σε ε, βαρβάρους κυριολεκτικά. Αυτό ας διορθωθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αυτά θα καταχωρηθούν στα πρακτικά και έτσι μπορείτε να ελέγξετε την αρχική διατύπωση και την απάντηση και την ανταπάντησή σας. Όλα αυτά θα έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά. Η κυρία Άννα Χέντεχερ παρακαλώ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου για την συγκέντρια κυρία Γκυόμ για την πολύ καλή και σκληρή δουλειά που έκανε στην έκθεση. Για, το... για τη δεύτερη φάση της ε, δέσμης μέτρων για το άσυλο. Πρόκειται για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ισχύσουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, αλλά ίδιε προδιαγραφέ, ελάχιστε τουλάχιστον προδιαγραφέ για το χειρισμό των ε, αιτήσεων ασύλου. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη όμω θα πρέπει να περιοριστούμε δηλαδή μόνο στα λόγια. Και αυτό είναι κάθε ολόκληρη τη Ευρώπη. Η Επιτροπή μας δηλώνει πως έχει την πρόθεση να καταθέσει νέα πρόταση η οποία θα προσεγγίσει περισσότερο τις ε, προτιμήσεις του Συμβουλίου, δυστυχώς. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε όμως τη σημασία αυτής της εκθέσεως και του σημαντικού μηνύματος που αποστέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι έχουν το δικαίωμα σε μία δίκη και εξέταση της αίτησής τους υπό δίκαιους όρους και κρίση της αιτήσεως ε, ασύλου κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, χωρίς βραθυπορίες και χωρίς επιπλέον δαπάνες. Είναι πολύ καλές ε, οι προτάσεις λοιπόν στην έκθεση. Θα ήθελα ιδιαίτερα όμως να υπογραμμίσω μία πρόταση τροπολογίας για εκείνους που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας όπως ανελικά παιδιά, αλλά και οι οικογένειες ε, που χρειάζονται κάποια καλύτερη υποδοχή. Ευχαριστώ Η κυρία Βίξτρομ ε, δεν είναι εδώ από ό,τι φαίνεται. Η κυρία Τάνια Φάγιομ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ την κυρία Γκυγιόμ, την εισηγητρία για την εξαιρετική δουλειά της. Χρειαζόμαστε ενοποιημένη διαδικασία για το άσυλο δίκαιη και ορθά λειτουργούσα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε παιδό, επί παραδείγματο η Μεσογείου. Χρειάζεται λοιπόν ένα κοινό σύστημα. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι ένα από τα κύρια ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόσφυγας ε, δεν θα πρέπει να τιμωρείται επειδή βρίσκεται στην κατάσταση αυτή και θα πρέπει ο στόχος μας να είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους στην διασφάλιση των βασικών τους ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βέβαια να βοηθούμε και τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ε, διεκπαιρέωση των ε, αιτήσεων. Δυστυχώ όμω ε, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είναι όλο και πιο πολύ η δυσπιστία με, την οποία τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες. Το βλέπουμε παραδείγματι στη Λαμπεντούσα την ζωφερή κατάσταση που αποδεικνύει ότι είναι ανεπιθύμητοι στην Ευρώπη οι πρόσφυγες. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από περιοχές κρίσης όπως ε, η Λιβύη για να βρουν ε, την ειρήνη, μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη αλλά και από άλλα μέρη της ε, Βόρειας Αφρικής θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια καλύτερη τύχη. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε θέση να υποδεχθούμε περισσότερους πρόσφυγες στο μέλλον με καλύτερες διαδικασίες ασύλου για δικό μας καλό αλλά και για καλό των ίδιων των προσφύγων. Αυτό ταυτόχρονα θα σημαίνει και λιγότερη επιβάρυνση των κρατών ε, που έχουν καλές επιδόσεις αυτή τη στιγμή με τον καταμερισμό του βάρους. Θα αποτρέψουμε επίσης τη μετατροπή της Ευρώπης σε ένα φρούριο και θα προσφέρουμε ασφαλή λιμένα σε αυτούς τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία Catch τώρα με τον κύριο Παπα-Νικολάου ως πρώτο One minute, please στα όσα υπόθηκαν θέλω και εγώ να συμφωνήσω ότι όλοι επιδιώκουμε αξιόπιστη και αποτελεσματική διαδικασία στην παροχή ασύλου και όλοι θέλουμε να περιφρουρήσουμε αυτούς τους σκοπούς. θα επικαλεστώ όμως και εγώ ένα παράδειγμα από την εμπειρία που είχαμε μερικούς μήνες πριν στην ελλάδα στην επίσημη αποστολή του κοινοβουλίου μας για τα θέματα ασύλου. όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο επισκεφτήκαμε το κέντρο κράτησης και εκεί ε, φιλοξενείται ένας υπήκοος τρίτης χώρας ε, στον οποίο ε, είχαμε ενώπιόν μας και συζητήσαμε μαζί του. Αφού λοιπόν μας είπε ότι είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, μετά από λίγο άρχισε να ομιλεί στα ελληνικά. Τον ρωτήσαμε λοιπόν πώς ήξερε ελληνικά και μας είπε, απήντησε, ότι ξέρω ελληνικά γιατί 10 χρόνια πριν εργαζόμουν στην Ελλάδα και είχα πάει τώρα στη χώρα μου και ξαναγύρισα και τώρα ετήθηκα άσυλο. Τι θέλω να πω με αυτό. Βεβαίω να τονίζουμε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές να περιφρουρήσουμε εκείνους που δικαιούνται άσυλο να προσέξουμε όμως και τι καταχρήσει. υπάρχουν διατάξεις που χρήζουν προσοχής αναφέρομαι και στις παρατηρήσει τη κυρίας χολμάιερ και κάνω κι εγώ μια επιπρόσθετη. λέμε ότι μετά από έξι μήνε το βάρο απόδειξη για εκείνον που διώκεται στην χώρα του μεταφέρεται στο κράτος μέλος και όχι στον ίδιο τον ετούντα. αυτό και μόνο δημιουργεί γραφειοκρατία και ίσως να είναι επιχείρημα για καταχρήσεις από κάποιους. σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκυγιόμ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Οι τροποποιήσεις ε, στην οδηγία όσον αφορά το άσυλο είναι ένα σημαντικό βήμα για να καταφέρουμε να θεσπίσουμε ένα κοινό σύστημα, κοινοτικό σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σαφήνεια των κανόνων και των διαδικασιών και διεργασιών είναι πρόσθετη, κύρια πρόσθετη αξία σε σχέση με αυτή τη νέα οδηγία. Θεσπίζονται διαφανείς κανόνες και κανονισμοί σε σχέση με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν έτσι να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα. Επίσης, διασφαλίζεται ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε αυτή την προστασία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διασφαλίζεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και είναι επίση σημαντικό να συνεχίσουμε με τη διαδικασία εναρμονισμού όσον αφορά τι εθνικέ νομοθεσίε για να αποφύγουμε παρεκκλήσει και διαφορέ μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων ασύλου που θα επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικό μα στόχο πρέπει να είναι η δημιουργία ενό πραγματικού κοινού συστήματο, κοινοτικού συστήματο ασύλου, όπω προβλέπεται από το πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Κύριε Πρόεδρε, όταν, αν υπάρχει κάποια βεβαιότητα είναι για το εξής. Τα επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτό μπορεί κανείς στις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων αλλά επίσης και στις εξελίξεις των τελευταίων ετών μπορεί να το καθορίσει κανείς εν μέρη όσον αφορά και τον τομέα του ασύλου αλλά και τη μετανάστευση ε, αντιμετωπίζουν υπερβολικές προκλήσεις και δεν τα καταφέρνουν μόνα τους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο πιστεύω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτά όλο και περισσότερες αρμοδιότητες και έτσι να μπορεί να δρά και να διασφαλίζει ώστε το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον να ρυθμίζεται από κοινέ αρχές και αξίες που θα είναι κοινέ για όλου. Ενιαίε προδιαγραφέ, δίκαιε διαδικασίε και διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά επίση από την άλλη πλευρά αποφυγή καταχρήσεων πρόληψη των καταχρήσεων. Είναι πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη ε, που συζητά, συζητείται πάρα πολύ έντονα. Αυτό είναι δύσκολη ε, πρόκληση και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η πρόταση οδηγίας για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας προκύπτει από το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν τελείως διαφορετικές εθνικές διαδικασίες ασύλου. Η Επιτροπή προσπαθεί να εναρμονίσει διαδικασίες και εργαλεία στον τομέα του ασύλου για να περιορίσει τις επανειλημμένες αιτήσει και προσφυγές. Κάποια κράτη στο Συμβούλιο ωστόσο δεν θέλουν να προχωρήσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τις απόψεις των κρατών μελών. Αν δεν ακούμε προσεκτικά αυτό που θέλουν να μας πούν τα κράτη, η δουλειά μας δεν θα είναι καρποφόρα. Ζητώ λοιπόν να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με τις αρχές των κρατών μελών της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συγκίτρια φοβάται προφανώς παρόλη αυτή, παρόλα αυτά τα κύματα προσφύγων από τη Βόρεια Αφρική λέει ότι δεν θα υπάρχουν ίσως αρκετοί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σε σχέση με το πριν ή μετά ε, και την επανένωση των ε, οικογενειών και ιδιαίτερη προστασία θα πρέπει να δίνεται σε άτομα, σε, πρόσφυγες, ε, με προβλήματα όσον αφορά την, ε, το φύλλο τους ε, ή την επιλογή τους, σεξουαλική τους επιλογή. Τώρα, σε σχέση με τις καταχρήσεις ε, ε, που σημειώνονται, είναι, ε, θα έλεγα, υπερβολικό να αναμένει κανείς ότι η ίδια αυτή η προσπάθεια θα καταβάλλεται από όλα τα κράτη-μέλη. Συναπατίζεται από διαφορετικά κράτη η Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης. Και σίγουρα, σε σχέση με ένα δημοκρατικό κράτος ένομης τάξης και δικαίου, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να καταχωρηθούν ως ασφαλή τρίτα κράτη ε, χώρες ε, για αυτά τα άτομα. Σας ευχαριστώ. Η διεθνής προστασία είναι ένας ε, κωδικός εφημισμός για το άσυλο που έχει χάσει τη δόξα του στο κοινό. Ωστόσο, οι αιτητές που περνούν από διάφορες ασφαλείς χώρες είναι μετανάστες κατ' επιλογή, όχι πρόσφυγες. Δεν έρχονται στην Ευρώπη Κάποιοι που έρχονται στην Ευρώπη από επισφαλείς χώρες μπορεί να είναι ατυχείς, αλλά δεν μπορούμε να, ε, να προστατεύσουμε ολόκληρο τον πληθυσμό πολλών χωρών. Η προστασία θα πρέπει να δίνεται στην πρώτη ασφαλή χώρα, εκεί όπου υπάρχει σχέση πολιτισμική ή ιστορική. Η Δύση και η Ευρώπη δεν θα πρέπει να γίνει χώρος υποδοχής όλων των ευάλωτων του κόσμου. Ο στόχος, μας θα, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να μειώσουμε την αστάθεια που οδηγεί στις μεγάλες μεταναστευτικές κινήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν πόλεμοι όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Πρέπει να φύγουμε από τη Λιβύη πριν οδηγηθούμε σε χερσαίο πόλεμο, να καταργήσουμε τις πιθανότητες πολέμου με το Ιράν και να ε, περιορίσουμε τις πιθανότητες Ιράξεων στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος, η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως πολλές φορές αναφέρθηκε, η συζήτηση για την οδηγία αυτή κρατά επί μακρόν. Από το 1999 είχαμε ως στόχο να υπάρξει μια κοινή πολιτική ασύλου. Τώρα υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο το 2012. Το αδιέξοδο που υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια αρχίζει και αλλάζει βλέπουμε το ξεκίνημα, το φως στην άκρη του τούνελ. Ευχαριστώ ιδίω το Κοινοβούλιο γιατί συνέβαλε σε αυτό. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα δίκαιο, αποτελεσματικό, συνεκτικό και ισοδύναμο σε όλα τα κράτη. Ήταν σαφές από το ξεκίνημα στις επαφές που είχαμε τους διάφορους εισηγητές για όλο το πακέτο μέτρων ότι θα έπρεπε να περάσουν κάποιες τροπολογίες, δεν είναι κάποιες αλλαγές, δεν είναι κάποια άποψη τη Επιτροπή αυτή. Είναι τέτοιο το αδιέξοδο που πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί, ώστε τα δύο σκέλη τη νομοθετική εξουσία να συμφωνήσουν. Και αύριο, η ψηφοφορία σα αύριο ή την Τετάρτη και οι προτάσει τη Επιτροπή νομίζω ότι επιτρέπουν να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε ένα πεδίο συμβιβασμού. Έχουμε έρθει σε επαφή με το Συμβούλιο όλη την Άνοιξη για να εντοπίσουμε τι βασικέ δυσκολίε. Αν θέλουμε να υπάρξει συμφωνία στο πακέτο ασύλου μέχρι το 2012 και να σα πω ότι σα σήμερα είναι τα 60 χρόνια τη σύμβαση τη Γενέβη και το λέω γιατί πρέπει να ε, ξεκινήσουμε κάποιου συμβιβασμού. Επαναλαμβάνω ότι το κείμενο αυτό είναι ο κρογωνιαίο λήθος όλου του ενιαίου συστήματος. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για τη δουλειά τους. Σε κυρία Γκυγιόμ. Δύο λεπτά. Oui, merci. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για όλες ή σχεδόν όλες τις παρεμβάσεις. Η κυρία κυρια χολμαιερ ε, απεχώρησε, αλλά θα τις μεταφέρει κάποιος, ότι δεν θα κουραστώ να, την, να προσπαθώ να την πείσω, ότι οι Τινήσοι θέλουν και μπορούν να τα καταφέρουν. Μια άλλη περίπτωση που θα πρέπει να εξετάσουμε επίση είναι ότι δεν θα πρέπει να ε, πιέσουμε τα κράτη-μέλη σε μια εναρμόνιση εκ των άνω αλλά μάλλον το αντίθετο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αντιδράσει και αντιρρήσει ή επιφυλάξει. Ε, αλλά από την άλλη θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν ότι αν οι πρωτοβάθμιε διαδικασίε είναι σωστέ και αποτελεσματικέ, θα κερδίσουν και εκείνα πολλά. Και ε, προ τα εκεί θα πρέπει να στραφούμε στου μεταρρυθμιστέ. Και άλλη μια τελευταία παρατήρηση. Ο ρόλο του Κοινοβουλίου είναι σημαντικό. Το ότι είμαστε συνομοθέτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλέ φορέ μα επεσήμανε πώ θα ήθελε ε, η γνώμη, η τοποθέτησή μας να έχει θεμελιώδη ρόλο για τη συνέχεια. Ε, ναι, λοιπόν, την Τετάρτη θα έχουμε την ευκαιρία ξεκάθαρα και απερίφραστα να ε, επιβεβαιώσουμε τις προτεραιότητες μας για μια εναρμονισμένη διαδικασία στον τομέα αυτών. Η συζήτηση έληξε, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Lightfried, έλεγχος των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίες διπλής χρήσης.